Pan Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε στις καρέκλες σας, καθίστε στις θέσεις σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu Κυρίσω την επανάληψη τη Συνόδου που διεκόπη στις 24 Μαρτίου του 2011. Τα πρακτικά της 23ης και 24ης Μαρτίου έχουν διανεμηθεί και ρωτώ εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ως προς τα πρακτικά. Άρα εγκρίνονται. Και θα ήθελα να προβώ σε μια σειρά ανακοινώσεων. Στις 26 Απριλίου θα χαιρετήσουμε, θα θυμηθούμε την 25η επέτειο από το Τσέρνομπιλ. Αποτείουμε λοιπόν, 25 χρόνια μετά, φόρο τιμής στα θύματα αυτής της καταστροφής, σε όσου έχασαν τη ζωή τους, σε όσους αγωνίζονται και ακόμη έχουν ορατά τα σημάδια αυτής της πυρηνικής καταστροφής. Οι αρμόδιες αρχές απέκρυψαν την καταστροφή αυτή από τις, ε, το λαό τους αλλά και από τις άλλες χώρες και εξ αυτού του λόγου κατέστη πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Το Τσέρνομπιλ στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε και αποτέλεσε και υπόδειγμα ε, συνεργασίας μεταξύ κρατών, μεταξύ, μέσα στη διεθνή κοινότητα. Καθώς λοιπόν ε, εορτάζουμε την 25η θλιβερή επέτειο του Τσερνόμπιλ, δεν μπορούμε να μην ε, στρέψουμε τα μάτια και το πνεύμα στο λαό της Ιαπωνίας, της Φουκουσίμα, σε εκείνου του ανθρώπους που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ξέρει ο σεισμός και το τσουνάμι. Δεύτερη πληροφορία. Πριν από ένα χρόνο στην περιοχή του Σμολένς και στις 10 Απριλίου συγκεκριμένα έχασαν τη ζωή τους μαζί με τον πρόεδρο της Πολωνίας 18 ε, λεφτές Πολωνοί και συνολικά 25 άτομα 96 ε, άτομα πολλοί ε, εκ των οποίων ήταν ε, εκπρόσωποι, αξιωματούχοι του κράτους της Πολωνίας. Πολλοί μάλιστα ήταν γνωστοί μου προσωπικοί. Ακόμη δεν είναι γνωστό το υπό ποιες συνθήκες έλαβε χώρα αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα. Περιμένουμε να λάβουμε τις τελικές πληροφορίες και αποτείουμε πάλι φόρο τιμής στους οικείους των θυμάτων, στα θύματα και στους οικείους τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εκφράζει την ανησυχία του για την απόρριψη από το Supreme Court των Δικαστήριων των Πολιτειών της προσφυγής του κυρίου Ντέιβις που ζητούσε αναβολή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής Με μία προσφυγή ο κύριος Τρόι Ντέιβις ζητούσε την μετατροπή της θανατικής αυτής ποινής από ε, θανατική σε ισόβια κάθεξη. Αυτό λοιπόν μας θλίβει βαθύτατα. Επίσης ανησυχούμε ιδιαίτερως για τις εξελίξεις στην αρχή του ελεφαντοστού. Οι προεδρικές εκλογές αντί να εξασφαλίσουν ειρήνη και ευημερία ε, ε, ρίξαν ε, τη χώρα στο χάος και την αναρχία. Ο Λογόν Μπακμπού δεν δέχθηκε την αναγνώριση της εκλογής του πολιτικού του αντιπάλου και έχει χρησιμοποιήσει κάθε είδου βία για να εξασφαλίσει την επικράτησή του στις εκλογές αυτές. Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι όποιο είναι υπέτειο για τέτοιου είδου πράξεις βία θα προσαχθεί στη δικαιοσύνη και σε αυτό θα συμβάλλει μεγάλη αυτή δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν τέλει, όπως σας είχα υποσχεθεί, πρέπει να δώσω ενημέρωση για ζητήματα διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Την Πέμπτη, λοιπόν, και ύστερα από μια συνεδρίαση της διασκέψης των Προέδρων, λάβατε μια επιστολή από πλευράς μου σχετική με το ζήτημα αυτό των κατηγοριών περί διαφθοράς εις βάρος ευρωβουλευτών. Λαμβάνουμε λοιπόν αποφασιστικά βήματα για την διατύπωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για τις ομάδες συμφερόντων και τις ομάδες πιέσεως, λόμπι, καθώς και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με το Προεδρείο, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα στι 6, για να συστήσει ακριβώς αυτό το θέμα και να λάβει αποφάσει για, την για περαιτέρω χειρισμού στην υπόθεση αυτή. Ο κύριος Νίκολσον έχει στήσει το λόγο στην θέση 603. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ στον φόνο την ε, Κυριακή στην Βόρεια Ιρλανδία ενός νεαρού αστυνομικού ο οποίος πήγαινε στη δουλειά